τον ε, αριθμό των αναφερομένων που ήρθαν στην ε, Επιτροπή Αναφορών για να παρακολουθήσουν ε, την πορεία των αναφορών τους. Είμαστε η Επιτροπή που έχει κατεξοχήν άμεσες επαφές με τους Ευρωπαίους πολίτες. Φάνηκε αυτό από τα στοιχεία με την παρουσία των αναφερομένων. Οπότε θα πρέπει να γίνουμε υπέρμαχοι των Ευρωπαίων πολιτών, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παστινάρο Κύριο Σαλαβράκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο την κυρία Βαλεάν για την εξαιρετική προσπάθεια που έχει κάνει και το ισορροπημένο κείμενο. Όταν μιλάμε βέβαια για ηθαγένεια μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερα. Και επειδή είμαι Έλλην την καταγωγή, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ξέρετε, εμεί οι Έλληνε έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία αναφέρεται ότι πάντων μέτρων είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό σήμερα, ε, διότι οι Λατίνοι πατριώτες σας κυρία Πρόεδρε είχαν πει κάτι άλλο. Homo hominis lupus. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος. Ε, δεν θα ήθελα να με σε αυτό, αλλά ήθελα να σας βάλω έναν γενικότερο προβληματισμό, κύριοι και κυρίες, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μιλάμε με συμπάθεια και δεν μπορεί διαφορετικά να μιλήσουμε, για, με συμπάθεια πάντα θα μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι ο ρόλος μας σαν πολιτικός και γι' αυτό ασχοληθήκαμε με την πολιτική για να βελτιώσουμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων, να αγαπάμε τους ανθρώπους Εκείνο όμως το οποίο βλέπω ότι πρέπει να δούμε και τους αριθμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, ε, είναι το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού και παράγει το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2030 οι στατιστικές λένε ότι ο πληθυσμός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι 4% και θα είμαστε το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δημιουργείται για την προσεχή 20 ετία ένα θέμα τεράστιου προβληματισμού μας. Και ο τεράστιος αυτός προβληματισμός έρχεται όχι μόνο από τη μείωση του πληθυσμού, αλλά και από το γεγονός ότι ενώ οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί σήμερα είναι 1 δισεκατομμύριο 600 περίπου εκατομμύρια παγκόσμια, το 2030 υπολογίζεται να είναι 2.200. 600 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι, δυναμικοί άνθρωποι, νέο αίμα, θα έρθουν στη γη, θα έρθουν στη ζωή τα προσεχή 20 χρόνια, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μία έχει μείωση πληθυσμού κατά 30 περίπου εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα ηθαγένεια και μετανάστευση που εν πολύ συνδυάζεται με την ηθαγένεια λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις. Πολλοί είμαστε εναντίον της ηθαγενείας, της παροχής ηθαγενείας σε ανθρώπους αλλοδαπούς ή παράνομους μετανάστες. Θα αναγκαστούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι πρωτού αναγκαστούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα στην προσεχή 20 ετία, να κανονίσουμε τους σωστούς κανόνες. Να βάλουμε σωστούς κανόνες εις τρόπον ώστε να μην μας ξεπεράσουν τα γεγονότα τα οποία φοβούμε ότι μας ξεπερνούν. Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι τα στοιχεία της εκθέσεως περιέχουν πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα τα υποστηρίξω και εγώ στην πολιτική μου ομάδα. Αλλά το θέμα μας είναι πάντοτε ε, να έχουμε στο νου και στην καρδιά μας ότι όσα λέμε και όσα πράττουμε και όσα νομοθετούμε ή όσα θέλουμε να νομοθετήσουμε πρέπει να είναι συνδυασμένα πιο κοντά με την πραγματικότητα. Και εκεί ε, φοβάμαι ότι το ψήφισμα, το οποίο είναι απόλυτα και νομικά και πολιτικά τέλειο, δεν θα έχει την εφαρμογή εκείνη την οποία θα πρέπει να έχει, διότι οι Λατίνοι έχετε δίκιο. Χόμο, hominis lupus. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Νεντελτσέβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με θερμές ευχαριστίες προς την εισηγήτρια για την ε, μεστή και εμπεριστατωμένη και πολύ διεξοδική της έκθεση για την ηθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει επιπλέον ε, εξουσίες και αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεκτημένο δεν αντικαθιστά βέβαια τις εθνικές νομοθεσίες, αλλά συμβάλλει και συμπληρώνει τις ε, ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμφωνώ με την κυρία Μπασέσκου για το σημείο 8. Στο σημείο 8 αναφέρεται ο περιορισμός της αγοράς εργασίας, ο περιορισμός, περιορισμός της πρόσβασης Ρουμάνων και Βουλγάρων πολιτών σε αγορές εργασίας. Και μέχρι τα 2000, το, το τέλη του 2011 οι χώρες μέλη έπρεπε να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ισχύουσες διατάξεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ενημερωθεί για την απόφαση ορισμένων χωρών να ανανεώσουν τους περιορισμούς της πρόσβασης ε, στις αγορές εργασίας μέχρι το 2013. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει εύλογος λόγος ε, για τον περιορισμό της πρόσβασης Ρουμάνων και Βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας ορισμένων χωρών μελών. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι η ελλειπής ε, ενημέρωση και η άγνοια πολλές φορές των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους να καταθέσουν αναφορές. Είναι πολύ σημαντικό να αφυπνίσουμε τους πολίτες, να διοργανώσουμε ενημερωτικές εκστρατείες και μέσω των εθνικών συνηγόρων του πολίτη για να βελτιωθεί αυτή η γνώση των Ευρωπαίων πολιτών ως προς το δικαίωμα αναφοράς. Γιατί δεν έχουν επίγνωση αυτού του μηχανισμού, παρόλο που είναι ανεκτήμητη σημασία για αυτούς. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην πρωτοβουλία, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, που θα λάβει σάρκα και οστά πολύ σύντομα. Καλό θα ήταν να ενημερωνόμαστε για την έμπρακτη εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών και να ενημερώνουμε και τους πολίτες. Ε, γιατί μας ενδιαφέρει η καθημερινότητά τους, η πραγματικότητα και όχι μόνο η θεωρία. Θεωρώ ότι η Ισπανία, η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι οι μόνες χώρες που αναφέρονται ως προβληματικές από την άποψη ε, κάποιων δικαιωμάτων ακινήτου περιουσίας, ε, διασυνοριακά ίδιος. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα και σε αλλα κρατημέλη και όχι μόνο στις τρεις χώρες που κατανομάζονται. Τέλος, ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Βαλεάν θερμά για την έκθεσή της και να τονίσω ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα, απτές δράσεις και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πιστεύω ότι αν συνενώσουμε τις προσπάθειές μας θα καταφέρουμε ε, να πετύχουμε. Πρόκειται για μια φετηρία, ένα ε, αρχικό βήμα, αλλά πολλά υποσχόμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ, κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαίρω και την κυρία Βαλεάν και κυρίως για την υπομονή που έδειξε, διότι περίμενε πάρα πολύ μέχρι να συζητηθεί επί της ουσίας αυτή η έκθεση, η οποία είναι εξαιρετική. Θα διαφωνήσω βέβαια με την προγνωμιλήτρια ως προς το ότι τα προβλήματα τα οποία είχαμε σε σχέση με τα δικαιώματα και δικαιώματα στην περιουσία ήταν ακριβώς σε χώρες αυτές που αναφέρατε, δηλαδή Βουλγαρία, Ισπανία και Κύπρο. Το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα τα οποία ε, τα βλέπουμε πανελειμμένα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, δεκάδες χιλιάδες αναφορές έχουμε λάβει για το θέμα αυτό. Το ίδιο και στην Κύπρο και στην Βουλγαρία. Σας συγχαίρω λοιπόν, διότι βλέπετε τα πραγματικά περιστατικά, ότι βιώνουν καθημερινά διακρίσεις πάρα πολλοί συμπολίτε μας. Δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό έτος ευρωπαϊκής ηθαγένειας καθημερινά. Κάθε μέρα θα έπρεπε να είναι η μέρα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Βλέπω και τη δική μου χώρα και χαίρομαι γιατί τονίζεται και τις διακρίσεις που υφίστανται κάποιοι και λόγω της θρησκείας που αυθαίρετα μπαίνει στην πολιτική συζήτηση άνθρωποι μιας διαφορετικής θρησκείας, μας διαφορετικής φυλής ή εθνικότητας, ε, φυλής, ε, φαίνεται να παρουσιάζονται ως πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο. Βλέποντας τα οικονομικά προβλήματα στην Ευρωζώνη, και δεν είναι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί μιλούσαμε για τον Ομένο Βασίλη, Είχαμε μια ε, έκθεση από το Migration Watch που ήταν αποτροπιαστική και η οποία έδειξε ε, βάσει μιας άλλης έκθεσης ότι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία της νεολαίας στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετίζονται άμεσα με τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των οποίων οι πολίτες δικαιούνται να πάνε να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπήρχε κάποιο επιχείρημα που να θεμελιώνει, που να τεκμηριώνει βέβαια αυτές, αυτούς τους ισχυρισμούς. Και ευτυχώς κάποιες ημέρες ε, μετά η κυβέρνηση αντέκρουσε ε, ε, ε, τα απορίσματα αυτής της έκθεσης. Υπάρχουν μέλη της κοινότητας των Ρωμά τα οποία απελάβνονται από την Ιταλία, από τη Γαλλία μόνο και μόνο γιατί θεωρούνται απειλή στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Τέτοια περιστατικά, τέτοια κρούσματα θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά στις χώρες μέλη μας εν καιρό που βλέπουμε ότι πολλοί καταφεύγουν σε πολύ κοντόθερο προστατευτισμό. Βλέπουμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα παραδείγματα. Ένα κράτο μέλο, το οποίο ήταν μέλο τη Ένωση για δεκαετίε. Πώ το επιτρέπει να πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να επιχειρηματολογεί για ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην μεσή διάταξη και μετά να ε, φεύγει λέγοντα ότι ε, τα προβλήματα τη υπόλοιπη Ένωση δεν με αφορούν. Μα όλα αυτά υπονομεύουν την ίδια τη βάση της, πάνω στην οποία δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ολοκληρώσω με το εξή. Το στένο το οποίο επιδείξατε ε, αντιμετωπίζοντα ζητήματα όπως η συνεχή άρνηση δικαιωμάτων σε ε, Βούλγαρους και Ρουμάνους πολίτες να μετεγκατασταθούν και να διαμένουν ελεύθερα σε διάφορες ε, άλλες χώρες, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χαίρομαι και είναι πολύ σωστό που το επισημαίνετε και το τονίζετε. Δεν μπορούμε να έχουμε μία κατηγορία ηθαγένες και μία ελαφρώς χαμηλότερη κατηγορία που δεν έχει τα ίδια δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει με ζευγάρια του ίδιου φίλου ή για τις διακρίσεις ε, που υφίστανται τα άτομα αυτά, τα οποία είτε είναι σε μια μόνη συμβίωση είτε έχουν νυμφευθεί και είναι του ίδιου φίλου. Δεν μπορούμε να στερούμε δικαιώματα από αυτού του ανθρώπου. Εσεί δείξατε σθένο. Όλοι οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν το ίδιο σθένο. Δηλαδή το σθένο να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που μπορεί να μην είναι δημοφιλή, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να επιληθούν εάν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα και να εξασφαλίσουμε την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε, είναι κάτι πολύ αόριστο και αφηρημένο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα γίνονται μόνο όταν μα αφορούν, όταν ε, θυγόμεθα εμεί. Τότε παίρνουν μια συγκεκριμένη μια ε, διάσταση απτή. Και αν έχουμε τη φαντασία και σκεφτούμε, ε, αν συνέβαινε αυτό σε μένα, αν συνέβαινε αυτό στην κόρη μου, στην ε, μητέρα μου, στον πατέρα μου, θα μου άρεσε, θα ήταν καλό. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, τότε δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό να συμβαίνει αυτό σε κάποιον άλλο, σε κάποιον τρίτο. Σας συγχαίρω λοιπόν που επιδείξετε αυτό το σθένος. Ίσως κάποια κράτη να μην θέλουν τις διαδικασίες παραβάση, να τις κινήσει δηλαδή η Κομισιόν, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτά τα κράτη ουσιαστικά κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια νομική βάση που συμφωνήσαμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Συγγνώμη που μακρηγορώ κυρία Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω. Κάποιε χώρε υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα, ή τα προβλήματα τη Ευρωζώνη, προκλήθηκαν από την υπερρύθμιση. Τα προβλήματα στην Ευρωζώνη πέραν των αγορών, των παγκόσμιων αγορών που έχουν αποφασίσει να κηρύξουν πόλεμο στι κυριαρχε χώρε τη Ευρωπαϊκής και στις οικονομίες μας. Τα προβλήματα τη Ευρωζώνη δημιουργήθηκαν επειδή ποτέ δεν τέθησαν σε εφαρμογή, δεν εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί. Εξού και είναι απόλυτο απαραίτητη έκθεση αυτή για να μα κατευθύνει, να μα δείξει που πρέπει να εστιάσουμε στην ε, Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα βασίζεται στο κράτο δικαίου και όχι στην απουσία νόμου. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι, κύριε Βαλεάν. Ε, Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στέκανε άλλο στο λόγο. Μπουλάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και στο συγγνώμη που καθυστέρησα τόσο. Κάποιος αποφάσισε να πέσει στις γραμμές του τρένου που με μετέφερε στις Βρυξέλλες και έτσι χρειάστηκε να αλλάξω δρομολόγιο. Για να έρθω να συστήσουμε αυτή την έκθεση ακριβώς που είναι τόσο σημαντική. Δεδομένων κυρίως των όσων έχει συμπεριλάβει στην έκθεση της κυρία Βαλεάν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διαβρύνουμε τη συζήτηση και πέραν του προβλήματος της διοικητικής αναγνώρισης, που δεν είναι αναγκαστικά η αναγνώριση του γάμου, αλλά η, δικαστική, η διοικητική αναγνώριση των ομοφιλοφιλικών ζευγών και βέβαια το πρόβλημα των Ρωμά, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η εκθέση ε, εν όλο για την ε, ηθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσο ευρύ το θέμα αυτό που θα κληθούμε πρώτα να ε, ενσκύψουμε σε άλλα προβλήματα και να τα διευρύνουμε. Λυπούμε λοιπόν που δεν ήρθα νωρίτερα και δεν άκουσα όλες τις παρεμβάσεις. Ε, σε μια προσπάθεια λοιπόν να αποφύγω τις ε, παναλήψεις θα περιοριστώ σε ολίγα αφού δεν ξέρω τι έχουν πει οι συνάδελφοι. Όλα λοιπόν τα προβλήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας που ευνοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα κενά, τα εμπόδια, τα οποία αντιμετωπίζει στην ελεύθερη του κυκλοφορία ο πολίτη, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, αναγνώριση επαγγελματικών ε, δεξιότητων και Θα πρέπει, Στέφα, να ε, υπογραμμίσουμε στην έκθεση αυτή την ανάγκη να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του ο πολίτης. Ήδη πολλά γίνονται, αν και μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα την κατάσταση. Και σημαντικό βρίσκω ότι όταν ενημερώνουμε τον πολίτη για τα δικαιώματα αυτά, θα πρέπει ταυτόχρονα να του επισημαίνουμε και τι δυνατότητες προσφυγής έχει για ε, να ε, αποκαταστήσει την περίπτωση όπου δεν εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα. Όπου λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει σωστή εφαρμογή των δικαιωμάτων ε, δεν υπάρχουν προβλήματα βεβαίως. Όταν όμως κάπου προκύψουν δυσκολίες στην αναγνώριση και την εφαρμογή, διαπιστώνω πάνω απ' όλα απουσία ενημέρωσης για τον πολίτη. Τι είδους ε, δικαιώματα έχει, τι προσφυγές και όλα αυτά. Τι ένδικα μέσα. Το ίδιο πιστεύω θα μας απασχολήσει τώρα με την, έκθεση, με την αναφορά για το Jugendamt, ότι υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης των νέων και γενικότερα του πολίτη ως προς τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να διεκδικήσει. Επίσης, ε, αυτή ο, ο συνδυασμός με, την, ε, ε, με το έτος 2013, έτος Ιθαγένειας δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι παρατηρήσεις κυρίας Βαλεάν μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες, πλην όμως περιορισμένες σε στενό κύκλο και θα πρέπει να τις διευρύνουμε. Η συζήτηση λοιπόν για την ηθαγένεια θα πρέπει να αναπτυχθεί και δει τώρα όπου μπορούμε πιστεύω και οφείλουμε να βοηθήσουμε τον πολίτη να ξεπεράσει την γραφειοκρατία, την ταλαιπωρία στη διοίκηση, το χρόνο και το χρήμα που δαπανά σε μια σειρά από διαβήματα προς τη δημόσια διοίκηση για κάτι το οποίο είναι ανεγνωρισμένο δικαίωμα. Κοιτάω λίγο και στα χαρτιά μου γιατί μπερδεύτηκα. Ναι, και έχω έρθει καθυστερημένα. Αυτά. Ε, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ. Ελα. Ο κύριος Μαρτίνες. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ κυρία Πρόεδρε την κυρία Βαλεάν για την έκθεσή της και να τη συγχαρώ γιατί πιστεύω ότι η προσπάθεια που έκανε ε, ήταν πραγματικά τιτάνια. Γιατί το να στάξει κανείς έκθεση για την ηθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι να θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει διδακτορική διατριβή, για να μην πω 20 διδακτορικές διατραβές. Πολύ δύσκολο λοιπόν το έργο της και το ε, και ανταπεξήλθε σε αυτό με πολύ ευφύ τρόπο, περιορίστηκε σε συγκεκριμένα και αυτά ζητήματα και όπως είπε και ο προλαλής σας, σίγουρα θα μπορούσαμε να τη διαβρύνουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αυτή την έκθεση, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ σωστή, αξιόλογη, ενδιαφέρουσα και δίνει τροφή και για συζήτηση. Και νομίζω ότι άλλο ατού της έκθεσης είναι ο ο δεύτερος τίτλος, να αρθούν ε, τα εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων ε, των πολιτών στην Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο τίτλος, ε, γιατί μας περιορίζει στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε εδώ, δηλαδή πώς θα τα εμπόδια που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών και όχι να συντάξουμε πραγματεία για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ας μην ξεχνούμε και την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013 και να συνδυάσουμε αυτό το θέμα με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Γιατί εκεί σε τελική ανάλυση θα βρούμε τα δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών και αυτό να το τονίσουμε όχι να είμαστε υπερβολικά διεξοδικοί και λεπτομεριακοί, αλλά να πούμε από τη στιγμή που έχουμε χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και μια και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσυπογράψει την Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήδη ανοίγουμε κατευθύνσεις πολύ πλούσιες και εκεί θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία θα διαπιστώσουμε ότι μένουν ανεκμετάλλευτα και δεν αξιοποιούνται πλήρως. Νομίζω ότι το τρέχον το 2012, θα μας δώσει μία μοναδική ευκαιρία για να επιχειρήσουμε και πάλι να αναθεωρήσουμε το πεδίο εφαρμογής των εργασιών μας την εμβέλεια των εργασιών μας. Γιατί είμαι εδώ και αρκετό καιρό δυσαρεστημένος με τον τρόπο λειτουργία μας. Όχι με το είδος του έργου που επιτελούμε, αλλά με τον τρόπο λειτουργία μας. Και νομίζω ότι ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλό εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών και την προσέγγιση των πολιτών, δυστυχώς έχουμε έχουμε μετατραπεί σε μία δομή ε, που λειτουργεί καλά, άσχημα, συγγνώμη, εσφαλμένα. Βέβαια, ο Αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο εδώ είναι κοινή ευθύνη, συλλογική ευθύνη, αλλά μερικές φορές ε, μετατρεπόμαστε σε ένα μηχανισμό που οδηγεί σε απογοήτευση και αμηχανία τους πολίτες που υποβάλλουν αναφορές. Αν δεν αποσαφινιστεί ότι εξετάζουμε αναφορές ή καταγγελίες για, για καταστρατήγηση ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ουσιαστικά μετατραπούμε σε ένα κουτί της Παδόρας που θα έρχεται ο καθένας και θα μας λέει το μακρύ του και το κοντό του, θα μπορεί να καταγγέλει οτιδήποτε, να μιλάει επί παντός επιστητού, είναι λογικό κάποιος ε, να έρχεται ε, σε μια εκλογική περιφέρεια και να συντάσει άρθρα με τίτλο η Ευρώπη δεν μας ακούει, η Ευρώπη κοφεύει και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη, αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει πολύ συγκεκριμένη λειτουργία, εξαιρετικά σημαντική αλλά συγκεκριμένη και που δυστυχώς δεν την αξιοποιούμε πλήρως, γιατί μερικές φορές αποσπά την προσοχή μας και χανόμαστε σε άλλα ζητήματα. Εγώ μίλησα με συμπολίτε μου που είπαν έχουμε κάνει την εξή καταγγελία και δεν ε, έλαβα απάντηση. Και συνέχεια βλέπουμε ε, ιδιαίτερα σε περιφερειακό τύπο ε, αρνητικές, ε, αρνητικές εντυπώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές και σε προγράμματα της τηλεόρασης. Λοιπόν, για το 2012 θα καλό θα ήταν να δώσουμε νέα έμφαση και να μπούμε στο σωστό δρόμο σε ό,τι αφορά το έργο της Επιτροπής και να αναφέρουμε, να κάνουμε μνήμα σημαντικών νομοθετικών κειμένων, όπως είναι ο Χάρτης Θεμελιών Δικαιωμάτων ή η Συνθήκη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αναφερόμαστε σε τέτοιου είδου κείμενα. Αυτά, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Καλή χρονιά σας εύχομαι και ευτυχισμένο το νέο έτος. Και φυσικά να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το έργο που επιτέλεσε μέχρι στιγμής η Πρόεδρος, αλλά και η Γραμματεία και η Δίκηση της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαρτίνες Μαρτίνες. Η έκθεση της κυρίας Βαλεάν αναφίβολα είναι αξιόλογη, όπως φάνηκε από τις ε, παρατηρήσεις που ακούσαμε. Θα της ξαναδώσω το λόγο για τα καταληκτικά σχόλια. Προηγουμένω όμω να υποβάλω και εγώ ορισμένε παρατηρήσει. Φυσικά θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ε, μεγάλη εκτίμησή μου και τον έπαινο μου προ την εισηγήτρια και την ικανοποίησή μου ως προς την πρόταση ε, πρωτοβουλίας για ένα τέτοιο θέμα που βρήκε σύμφωνος τους συναδέλφους της Επιτροπής. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Μαρτίνες Μαρτίνες ότι είναι σημαντικό το δεύτερο τμήμα του τίτλου ε, της έκθεσης που μιλάει για άριστον εμποδίο στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι πολύ σωστά οριοθετούμε το περιεχόμενο της έκθεσης και φυσικά ε, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το έργο της Επιτροπής ε, που είναι να προβάλλουμε καταγγελίες για παραβίαση της ε, εθνικής νομοθεσίας. Η κυρία Βαλεάν εντόπισε κάποια εμπόδια σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών και υπέβαλε προτάσεις για την άρση αυτών των εμποδίων προκειμένου να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ελπίζω τις επόμενες μέρες που θα ξανασυζητήσω το θέμα με την κυρία Βαλεάν, να μπορέσω να καταλήξω σε κάποιες τροπολογίες για να συμβάλλω και εγώ στη διαμόρφωση της έκθεσής της. Μετά την παρέμβαση του κυρίου Κάσμαν, ε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή Αναφορών να επιτελεί το έργο και τη λειτουργία της, που είναι η έμπρακτη προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια πιο αυστηρή εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είπε ο κύριος Μαρτίνες. Προσοχή όμως, δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της σύγχυσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τα δικαιώματα του πολίτη. Γιατί Αυτά τα πολιτικά δικαιώματα εμπίπτουν στη νομική βάση και τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε γιατί δεν ισχύουν παντού αρμοδιότητες. Καλό θα ήταν λοιπόν να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Και επίσης και για τα δικαίωμα παραμονής ε, είναι σημαντικό αυτό το θέμα και γνωρίζουμε ότι υπάρχει οριοθετωμένη αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, την ε, επιμέλεια των παιδιών, ε, διαζύγια, αναγνώριση ζευγαριών του ίδιου φύλου. Αν και στην περίπτωση αυτή ίσως δεν εμπίπτουμε ε, στην εθνική αρμοδιότητα, ε, δεν θα πρέπει να επισέλθουμε μάλλον στην εθνική αρμοδιότητα. Απλώς ε, θα πρέπει κάποια εμπόδια να, να τα άρουμε για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους που απορρέουν από την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο σημείο που καλό θα να το αναφέρουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό είναι οι διαφημίσεις για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Ε, το επισήμανε αυτό κυρία Βαλεάν. Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διδάσκαλοι ξένων γλωσσών και ίσως αυτό το θέμα ε, δεν περιοριστεί μόνο στη συγκεκριμένη αναφορά που περιλαμβάνει κάποιες καταγγελίες, αλλά ε, μπορούμε να το δούμε και πιο γενικά. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε αρκετά συχνά. Οπότε καλό θα ήταν να το εξετάσουμε. Και τέλος... τα, η άσκηση των, δικαιωμάτων, των περιουσιακών δικαιωμάτων στην Βουλγαρία, Ισπανία και Κύπρο. Για τα θέματα αυτά θα πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα τι είδους παρέμβαση θέλουμε από την Επιτροπή, ώστε να μην ε, ε, προσκρούσουμε στην ε, κατηγορηματική απάντηση ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα. Έχουμε πολύ συχνά αναφορέ για παραβίαση των περιουσιακών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα από αυτέ τι τρει χώρε. Και υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να δούμε α, οι παρεμβάσει μα να, ε, να οριοθετηθούν από τι αρμοδιότητέ μα. Αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια την κυρία Βαλέαν και να σας υπενθυμίσω και τη διορία για την κατάθεση των τροπολογιών που λήγει στις 19 Ιανουαρίου. Η έκθεση Βαλεάν θα ψηφιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής που θα λάβει χώρα στις 27 Φεβρουαρίου ώστε να περάσει στην μήνυ ολομέλεια του Μαρτίου. Δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο που προβλέπει την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013. Θα γίνει παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εκπρόσωπο μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Σοφή Μπερνάρ και λυπούμε αν κατακρεούργησα το όνομά της. Thank you very much. Hello, ladies. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Σοφή Μπεχνάχ είναι το όνομά μου και είμαι επικεφαλής της ομάδας για την πολιτική ε, για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να σας παρουσιάσω αυτή τη γνωμοδότηση για την Ευρώπη την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια καλύτερα το 2013. Ξέρετε ότι θα λάβει χώρα μέσα σε πολύ σημαντικό χρονικό πλαίσιο αυτή η χρονιά, ένα χρόνο δηλαδή πριν από τις ευρωεκλογές του 2014 και επίσης με την, ε, και λίγο πριν την εισαγωγή της ε, Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας που θεσπίζει η συνθήκη του Μάστριχτ. Επίσης δεν θέλω να πω λοιπόν ότι διαπιστώνεται πως χρειάζονται όλο και περισσότερες προσπάθειες να, να ενθαρρύνουμε τους ε, πολίτες για να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Για μας την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, μεγάλο καθήκον είναι να εξηγήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες και λύσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Θα θυμάστε ασφαλώς ότι το Δεκέμβριο του 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Χρονιά έτσι ώστε να δώσει νέα όθηση στη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και να ενημερωθούν ε, οι, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πολίτη τον αληθινό άνθρωπο δηλαδή. Οι περισσότεροι βέβαια στην ερώτηση αυτή απαντούν λέγοντας ότι είναι η ελευθερία ταξιδιού ή σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων είναι αυτό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι είναι δεδομένο δικαίωμα, ε, συνυφασμένο με την Ευρωπαϊκή ηθαγένεια το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση, στην ελεύθερη κίνηση. Ε, και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό ακριβώς ε, το χαρακτηριστικό αυτό δεδομένο για να υπογραμμίσουμε την έννοια της Ευρωπαϊκής Ταγένειας και να εξηγήσουμε καλύτερα στον πολίτη τι σημαίνει στην πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, λογικό και απαραίτητο το προσεχές βήμα που θα προτείνω να ενημερώσουμε τον πολίτη, να τον ευαισθητοποιήσουμε για τα δικαιώματά του στην ελεύθερη διακίνηση, πράγμα το οποίο πιστεύω θα επιτρέψει στον πολίτη και να ασκεί καλύτερα τα δικαιώματά του να κινείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει καλύτερη αίσθηση του ανήκει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενστερνιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν αυτού όμως δεν περιορίζεται μόνο στην ευαισθητοποίηση Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να προξενήσουμε συζήτηση, διάλογο για τα ε, ωφέλη της ε, ελεύθερης ε, διακίνωσης, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής δηλαδή και αμοιβαία κατανόηση και γνώση του πολίτη των πολιτών μεταξύ τους οι βασικές αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το πνεύμα αποδοχής, η αλληλεγγύη, η διαλλακτικότητα πρέπει νομίζω να υπογραμμιστούν ιδιαίτερως εναντί των κινδύνων των ε, ε, ακροτήτων του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει τις σχετικές προσπάθειες βεβαίως σε κεντρικό επίπεδο, αλλά αναμένει και ότι θα αναπτυχθούν αντίστοιχα αποκεντρωμένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσεως τοπικό επίπεδο ε, που θα στηρίξουν τις κεντρικές προσπάθειες της Επιτροπής. Πρέπει όλες να εργαστούμε, Δηλαδή, η στρατηγική εταίρη τη εκστρατείας θα είναι βεβαίω όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη-μέλη, θα διαδραματίσουν κέριο ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εκστρατεία, οι εθνικέ κυβερνήσει, αλλά και οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών με τη δικτύωσή του ε, θα συμμετάσχουν επίση πλήρω και έχουμε ήδη ξεκινήσει επαφέ μαζί του. Οι υπηρεσίε επιτροπή στο σύνολό του, με ιδιαίτερα η έμφαση βέβαια στι εκείνε που έχουν σχέση με τον πολίτη πολίτη θα κληθούν να αναπτύξουν μέσα στο πλαίσιο των δικών τους πόρων ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Το ευρωπαϊκό έτος αυτό λοιπόν θα στρέφεται και θα απευθύνεται στο γενικό κοινό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η εκστρατεία θα πρέπει να στηριχθεί σε παράγοντα πολλαπλασιαστικό για να απευθύνει το μήνυμα την πληροφορία όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο κοινό ε, πιθανοί τρόποι δράσης και πρωτοβουλίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό, τοπικό, περιφερειακό επίπεδο βεβαίω μπορεί να ε, αναπτυχθούν παραδείγματι εκστρατείες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, κοινέ ε, πρακτικές και ενημέρωση για κοινέ πρακτικές, ευρύτερος διάλογος, συζητήσεις. Επέραν αυτών όμως ε, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε και το ρόλο του U-Direct και του Europe ε, τα δύο αυτά πορτάλ δηλαδή που αποτελούν εργαλεία του συστήματος ενημέρωσης για τα δικαιώματα του πολίτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, συνεργαστούν κατά τρόπο στρατηγικό για να μετατρέψουν αυτό το ευρωπαϊκό έτος σε μια επιτυχή χρονιά. Θα ήθελα λοιπόν ε, με κάθε ευκαιρία να συστήσουμε τις προτάσεις μας και βεβαίω να δώσω απαντήσεις οποιαδήποτε απορία ενδεχομένως έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι μπορεί τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση για το έγγραφο αυτό. Που σχετίζεται βέβαια και με την έκθεση του κύριου Σαλαβράκου, στον οποίο δίνω πρώτο το λόγο. Ε, επαναλαμβάνω ότι η παρουσίαση από πλευρά της Επιτροπής νομίζω και αρκετά φιλόδοξη διότι παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής αποτελεί ένα μέρος του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αναπτύχθηκε από το παράγωγο δίκαιο, από τις ε, ε, τοπικές νομοθεσίες, οι πολίτες της Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε άλλα κράτη-μέλη. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 2010 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποτελεσματική εφαρμογή μετά την έναρξη της ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διαθέσει το 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος για την Ιθαγένεια. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση για την Ιθαγένεια του 2010 η Επιτροπή πολύ σωστά προσδιορίσε και αποδεικνύεται με παραδείγματα από την πραγματικότητα τα εμπόδια που οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, των δικαιωμάτων ως πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον η Επιτροπή έχει υποδείξει νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, με, οι οποίες μαζί με το έτος της πρότασης για τα υπάρχοντα κενά θα πρέπει να βελτιώσουν την εν γέννη κατάσταση. Μία από τις προτάσεις είναι να επιτρέψει τόσο τους απλούς πολίτες όσο και στους νομικούς να βρίσκουν εύκολα πολυγλωσσικές πληροφορίες για τη δικαιοσύνη μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και να ενημερώνονται το συνομότερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένου ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ένα από τα πιο εύκολα και προσβάσιμα μέσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει κατά την άποψή μου στεναρά αυτή την ιδέα. Από πλευρά μου θεωρώ ότι πρέπει να θέσουμε τους εξή κατά βάση στόχους. Πρώτον, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων να είναι αναφέρετο δικαίωμα των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματο των πολιτών, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν στο κράτος μέλο τις αρεσκίες τους. Δεύτερον, έχει ζωτική σημασία να ενημερώνονται σωστά οι πολίτες για τα δικαιώματά τους όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλο κράτος ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει η διασφάλιση ή η δυνατότητα διασφάλισης ομαλούς διαβίωσης. Τόσο ε, σαν διαβίωση όσο σαν ε, και επαγγελματική εξέλιξη. Τρίτον, οι εργαζόμενοι που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια κράτους μέλους και εφόσον είναι νόμιμο πολίτες να τους παρέχονται τα ίδια δικαιώματα με αυτά που παρέχονται στους πολίτες που ζουν σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικό προβληματισμό είχα αναπτύξει και προηγούμενα όταν αναφερόμουν στην έκθεση της κυρίας Βαλέν. Και τέταρτο θεωρώ ότι το δίκτυο EURES πρέπει να αποτελέσει όχημα διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες εργασίας σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στη συγκεκριμένη περίοδο που η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την ανεργία. Ε, με ιδιαίτερη χαρά θα δεχθώ υποδείξεις και συμπληρώσεις των συναδέλφων, ώστε το κείμενο να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και θα είναι τιμή μου να ε, ενώσουν τις σκέψεις τους μαζί μου, να βελτιώσουμε την κατάσταση και να βγάλουμε κάτι το καλύτερο και με την Επιτροπή βεβαίως ε, διαβεβαιώ ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα σημεία αυτά βεβαίως σχετίζονται άμεσα και με τα θέματα που συζητήσαμε νωρίτερα, την ηθαγένεια βεβαίω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για μένα το έτος του Ευρωπαίου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ιταγένειας είναι πάνω απ' όλα μια προβολή εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε και ο συνάδελφο, πρέπει να ενημερώσουμε τον πολίτη για τα δικαιώματά του. Αυτή είναι η πρόθεση τελευταία ανάλυση, ο τελικό σκοπό ε, το, ο πυρήνα όλη αυτή τη υπόθεση. Και γι' αυτό θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω πολύ για την πρωτοβουλία και δεύτερον να συμπληρώσω και, για το και σε σχέση με το προηγούμενο σημείο στην Μερσία. διάταξη. Μπορεί να έχουμε πολλέ διαφωνίε. Μπορεί, Φερρυπίν, ε, σε μια ενδεχόμενη δημοσκόπηση, οι πολίτες να μα έδειχναν ότι δεν ξέρουν ακριβώ τι σημαίνει πολίτης Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Αλλά στην πράξη το ξέρουν. Μπορεί θεωρητικά να μην το ξέρουν στην πράξη, όμω το ξέρουν. Και το βλέπουμε αυτό και με τις πολυάριθμε αναφορέ που έρχονται. Ότι ο πολίτης όταν διαπιστώνει ότι μα χρειάζεται, ναι, διεκδικεί. Διεκδικεί και διεκδικεί και την ε, ελεύθερη διακίνηση, το δικαίωμα στην κυκλοφορία. Ε, άρα περισσότερο το θέμα μας είναι ίσως η ασφάλεια δικαίου, όπως θα μπορούσα να το περιγράψω, Δηλαδή το να μπορεί, εάν κάποιο έχει ε, μετακομίσει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και μετά του έρθει μια κληρονομιά από το προηγούμενο κράτος μέλος, να μην έχει πρόβλημα ω προ τα ε, δικαιικά πλαίσια στα οποία θα κινηθεί, θα, θα αναπτυχθεί αυτή η διαδικασία τη κληρονομιά. Αυτό θα είναι περισσότερο το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στον πολίτη πολύ ξεκάθαρο ότι έχει δικαίωμα, έχει δικαίωμα σε προσφυγή για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς ο σκοπός και το νόημα του Ευρωπαϊκού Έτος. Επίση, από πλευρά ε, τη Επιτροπή των Αναφορών, θα ήθελα να επισημάνω ότι εάν διαπιστώνεται κάποια έλλειψη στη δική μα δουλειά, την έλλειψη εγώ αυτή θα την εντόπισα περισσότερο σε ένα σημείο. Ότι διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο έλλειμμα, κάποιο πρόβλημα, ενημερώνουμε και τον ετούμενο, Φερρυπίν, για τα δικαιώματα, τα πολιτικά του δικαιώματα, ποια είναι, αλλά δεν έχουμε αρκετά δημοκρατικά, κοινοβουλευτικά μέσα για να επιβάλλουμε την ουσιαστική υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν θα έλεγα και απευθυνόμενος και προς τους φίλους μας και στις άλλες επιτροπές. Όταν, μπορούμε, όταν διαπιστώσουμε μια τέτοια έλλειψη, ένα κενό, ως κοινοβούλιο να αναλαμβάνουμε δράση για να διεκδικήσουμε και να επιβάλλουμε την αποκατάσταση ε, του δικαίου γιατί βεβαίω υπάρχει η ευρωπαϊκή διάσταση και πέραν των τοπικών ή περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων θα πρέπει να είμαστε σε θέση και να συζητούμε όπου υπάρχουν τέτοιε διαφορέ, και να οδηγούμαστε προ ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα με την επιλογή μα. Και επίσης Προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν θέλουμε να έχει μόνο κεντρική οργάνωση αυτό το ευρωπαϊκό Έτο. Δεν θέλουμε μόνο οι Βρυξέλλες δηλαδή να, κάνουν την επικοινωνιακή, να έχουν την επικοινωνιακή πρωτοβουλία. Θέλουμε να υπάρχουν και οι περιφερειακές πτυχές. Θέλουμε να υπογραμμιστεί το, το έτος αυτό ως έτος που θα ανήκει στις περιφέρειες και γι' αυτό ρωτάω Υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχουν κλήσεις προς τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε κάποιες πρωτοβουλίες. Γιατί βεβαίως πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει τα δικαιώματά του για να τα διεκδικήσει και όταν τα γνωρίζει μερικές φορές εντοπίζει και κάποιου προβλήματα ή ελλείψεις και έτσι πρέπει κάπου να απευθυνθεί, να μπορεί να απευθυνθεί για να, αποκατασταθεί ή, ε, να αποκατασταθούν τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ. Νεβέλτσεβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα ε, δρατώμενη τη ευκαιρία να ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαίρετη αυτή πρωτοβουλία. Είναι προφανές και για μας ότι όλο αυτό το θέμα έχει άμεση διασύνδεση με τα ζητήματα που μας απασχόλησαν μόλις τώρα. Με χαρά λοιπόν διαπιστώνουμε ότι επιτέλους αναγνωρίζεται ένα ευρωπαϊκό έτος αφιερωμένο στον πολίτη. Από την έναρξη αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος οι κύριες πρόοδοι σημειώνονταν και σημειώνονται όταν ο πολίτης τίθεται στο επίκεντρο της Ευρώπης. Και εδώ ακριβώς είναι και το κύριο εμπόδιο που θα πρέπει να αντιπαρέλθουμε. Το να θέσουμε τον πολίτη στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι αυτόματα υποχρεούται και να βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν πρέπει να εντοπίσουμε τις διαφορές μεταξύ της μακράς ιστορίας που έχει πλέον το ευρωπαϊκό ολοκλήρωμα και της ε, άγνοιας σε μεγάλο βαθμό του πολίτη για τα δικαιώματά του. Αυτή είναι η κύρια πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η κύρια πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε ώστε η τάφρο αυτή που πολλέ φορέ υπάρχει μεταξύ του νομικού πλέγματο που έχει ε, εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη γνώση του πολίτη για τα δικαιώματά του να κλείσει σιγά σιγά. Το έτο αυτό, το Ευρωπαϊκό Έτο για τον Πολίτη του 2013 θα σημάνει λοιπόν την αποστολή ενό μηνύματος ότι έρονται όλα τα εμπόδια, εφαρμόζεται πλήρω η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Επίση, το μήνυμα αυτό θα σημαίνει και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση γιατί μπορεί να έχουν περάσει 20 χρόνια αλλά αυτό ταυτόχρονα σημαίνει και ενηλικίωση σημαίνει και ορίμανση, σημαίνει και περισσότερο πλουραλισμό και άρα χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες δράσεις. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη εγκύτητα του πολίτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με το δικαίωμα να προασπίσετε τα δικαιώματά του και ταυτόχρονα με την αίσθηση ότι βλέπει συγκεκριμένες δράσεις στην καθημερινότητά του βλέπει να υλοποιείται στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι πιστεύω ότι με τη θέση εφαρμογή, σε ισχύ μάλλον Συνδική Λισαβόνα, βεβαίω σημειώνονται κάποιε πρόοδοι. Φερρυπίν στη δικαιοσύνη. Θυμάμαι στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών τη χαρά που είχαμε εκφράσει όλοι μα όταν ανατέθηκαν νέε εξουσίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούσαμε πλέον να διεκδικήσουμε το δικαίωμα για τη μετάφραση. Επίση όμω θα πρέπει να αγωνιζόμαστε και για καλύτερη ενημέρωση για τη δικονομία, για του δικονομικού και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Σιγητή, με τον κύριο Στάκτη τη Κομοδότηση, όταν επισημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβαση σε πολύγλωσσε υπηρεσίε ενημέρωση για τη δικαιοσύνη μέσω του e-justice, του ευρωπαϊκού αυτού πόρταλ που δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε. Επίση θα πρέπει να συνεχίσουμε να προβάλλουμε τα δικαιώματα των πολιτών ω καταναλωτών τουριστών, επισκεπτών, ε, επιβατών σε μέσα μαζικής, ε, μαζικών μεταφορών και γι' αυτό το πρώτο μου ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν ποιε συγκεκριμένε πρωτοβουλίες έχετε υπόψη για τον τομέα αυτό και υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαμε εμείς οι ευρωβουλευτές να έχουμε υπόψη για να μπορέσουμε να διαδώσουμε και να ε, εκλεγεύσουμε τροποντινά αυτή τη γνώση, αυτά τα στοιχεία προς τον Ευρωπαίο πολίτη. Επίσης θα θέλω να πω ότι μια τέτοια χρονιά δεν μπορεί να επιτύχει και κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς συμμετοχή των νέων. Η επιτυχία δε του μεγάλου προγράμματος έρασμου απέδειξε πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι νέοι στην κουλτούρα, στον πολιτισμό και συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια. Η ε, αναγνώριση λοιπόν διπλωμάτων ε, και δεξιοτήτων, επαγγελματικών δεξιοτήτων αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα για τους νέους πολίτες της Ευρώπης ήθελα να ρωτήσω ποιε είναι οι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε στο τομέα αυτό και όταν μιλούμε για την ε, ημέρα αυτή, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για οργάνωση με συνεκτικό τρόπο των πρωτοβουλειών που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Ιθαγένειας και συγκεκριμένα τις δράσεις ε, και ε, νεολαία εν κινήσει. Όχι νεολαία εν δράση, το καινούριο πρόγραμμα νεολαία εν κινήσει που πιστεύω θα μπορούσε να αποτελέσει ταυτόχρονα και μια νέα εγγύηση για να αντιμετωπιστούν ή να ε, παραμεριστούν τα εμπόδια που ενδεχομένω αντιμετωπίζουν οι νέοι. Φυσικά θα επανέλθω και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην ελεύθερη διακίνηση. Είναι κάτι που μα απασχόλησε και νωρίτερα, γιατί πώ μπορούμε να εξηγήσουμε στον ε, Βούλγαρο και τον Ρουμάνο εργαζόμενο ότι δεν έχει πλήρη ελευθερία κίνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκατάσταση για να εργάζεται. Αυτό λοιπόν και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για πλήρη δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν τον Ευρωπαίο πολίτη ως προς τα δικαιώματά του θα πρέπει να καταγραφούν έτσι ώστε πράγματι να ανταποκρίνονται στι στις ανάγκες του πολίτη. Δηλαδή ε, καλό θα είναι οποιαδήποτε εκδήλωση να μην είναι μια εκδήλωση μέσα από την οποία απλώ εμεί θα εκφράζουμε τι ε, προθέσει μα ή τι ευχέ μα, γιατί μπορεί να μην ε, ταυτίζεται αυτή με τι ανάγκε του πολίτη. Θα πρέπει για να υπάρχει αυτή η αναγνώριση, αυτή η ταύτιση, να περνάμε μέσα από το σωστό εργαλείο που είναι η γλώσσα, η επικοινωνία δηλαδή και με συγκεκριμένε δράσει και πρωτοβουλίε να συνεχίσουμε να προβάλλουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με ένα κάπω λυρικό ύφο, αλλά χρειάζεται και λίγη γλύκα σε αυτό τον τόσο σκληρό και άπονο κόσμο, όπως λέμε συχνά, σε αυτό το ευρωπαϊκό Έτο των πολιτών σε... και χάρη και σε αυτή την έκθεση που μόλι συζητήσαμε, πρέπει πιστεύω επιτέλους να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, να την απαλλάξουμε καλύτερα από το καβούκι ε, και το βαρύδι που αποτελεί μερικές φορές ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και να την καταστήσουμε ένα πραγματικό ζώντα οργανισμό του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω κι εγώ συμπληρωματικά και αυτό το ευρωπαϊκό έτος σε σχέση με το όσο είπε ο κύριος Γιάρ τα εξή. Συμπληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι και το τοπικό και το εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συμπεριληφθούν Και αυτό δεν θα το εξασφαλίσει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο με κάποιες εκστρατείες. Γιατί ναι, βεβαίω πρέπει να υπάρχει η κεντρική οργάνωση τη εκστρατεία, αλλά απαραίτητο είναι να υπάρξει και η οργάνωση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και θα ήθελα επίση να συμπληρώσω με εξή. Ότι υπάρχει βεβαίω η πρωτοβουλία και η ιδέα μέσα στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά υπάρχει και η άλλη πτυχή, που είναι η πτυχή τη κοινωνία των πολιτών μη κυβερνητικές οργανώσεις και μη επίσημες οργανώσεις, άλλες μη επίσημες οργανώσεις που θα πρέπει να συμμετάσχουν, να συνδεθούν σε αυτήν την πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Έτος, το οποίο πρέπει από κοινού με την κοινωνία των πολιτών να αναπτυχθεί και να σχηματιστεί, να διαμορφωθεί. Επίσης, Πιστεύω ότι αυτή η διάσταση κοινωνία των πολιτών δηλαδή ιδιαίτερα μπορεί να προσφέρει τα μάλα ως προς την επικοινωνία. Επικοινωνιακή πολιτική την οποία θα ήθελα να προσδιορίσω ως εξή και με πολύ στενό ε, με πολύ σταλτικό τρόπο. Εάν έχουμε μια κεντρική εκδήλωση της Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου ε, φέτος, αυτό το έτος μάλλον, δεν θα είναι επικοινωνία στο βαθμό που κανείς δεν θα γνωρίζει ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή εκδήλωση για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, εκτός από αυτούς που έχουν προσκληθεί και πάνε εκεί. Εάν όμως από την άλλη υπάρξει μια ιστοσελίδα, που πάλι δεν αρκεί, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να ενδιαφερθεί κάποιος να κοιτάξει στο Google και να καταλήξει τη σελίδα αυτή. Άρα πάλι δεν ε, είμαστε στο επίπεδο που απαιτούν οι περιστάσεις και οι χρονιά αυτή. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι, θα έλεγα σχεδόν επιθετικοί. Χρειάζεται μια επαγγελματική και με τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα ε, ανάπτυξη, επικοινωνία και λυπούμε που είναι τόσο ελλειπής, που ήταν μάλλον τόσο ελλειπής η χρηματοδότηση του έτους εθελοντισμού και του έτους ε, δραστήριων γερατιών, θα έλεγα ίσως όχι επονίδιστη για την ευαριά κουβέντα, αλλά πάντως λυπούμε πάρα πολύ που τελικά με 500 μόλις εκατομμύρια ευρώ θελήσαμε τάχα να απευθυνθούμε στον Ευρωπαίο πολίτη και θεωρήσαμε ότι έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η προσέγγιση, είναι καλή η ιδέα της χρονιάς, ανεξαρτήτως όμως των όποιων των επιφυλάξεων προβληματισμών έχουμε λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν διαθέτουμε αρκετά κονδύλια. Πρέπει λοιπόν το ταχύτερο δυνατό να περάσουμε στον, ε, στη δουλειά που έχει να κάνει με το σχεδιασμό και με την ανάπτυξη στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Χρονιά. Ευχαριστώ. Γιώτοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι συζητούμε τα δικαιώματα των πολιτών ε, για δύο ώρες περίπου, συζητάμε διάφορες πρωτοβουλίες, διάφορες εκθέσεις. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση αυτή πηγαίνει προς μια κατεύθυνση που δεν φαίνεται να είναι και τόσο επικοδομητική. Δηλαδή, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει κάποια διάρθρωση πάνω σε αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε. και σε ό,τι αφορά το μελλοντικό μας έργο προς τους ε, πολίτες. Ακούστε λοιπόν τι θέλω εγώ να προτείνω, αλλά πρώτα μια ερώτηση. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα έγγραφο ή θα υπάρξει ένα έγγραφο που μπορούμε να μελετήσουμε και να συζητήσουμε και επί του οποίου να υποβάλουμε ενδεχομένω προτάσεις, δηλαδή μια εκστρατεία στα διάφορα κράτη-μέλη, χρήσιμο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Κάθε χρόνο, κάθε έτος είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα. και καλό θα ήταν κατά την άποψή μου, αν είναι δυνατόν βέβαια, να ε, συζητήσουμε κάποια στιγμή στην Επιτροπή μας ε, πόσο αποτελεσματικές κρίνει τις διάφορες εκστρατείες η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος, η Κομισιόν θέλει να απαντήσει τώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Θα απαντήσω στα ερωτήματα. Αρχίζοντας από την τοπική περιφερειακή εθνική διάσταση. Είναι προφανές ότι θέλουμε φυσικά να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, να συνεργαστούμε με τις περιφέρειες. Αύριο έχουμε και μια συνεδρίαση με την Επιτροπή των Περιφερειών ε, και θα δούμε και με τις ε, τοπικές ε, κοινότητες και τις κοινότητες Ευρώπης τις επόμενες ημέρες, ε, τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού και η κοινωνία των πολιτών. Έχουμε έναν άτυπο, μια άτυπη συμμαχία, αν θέλετε, ή συνασπισμό με διάφορες οργανώσεις που διαμορφώνεται σιγά σιγά και θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους αυτούς τους οργανισμούς, να ακούσουμε τις προσδοκίες τους, ε, τα αιτήματά τους, τις προτάσεις τους. Σίγουρα ισχύει και η ΕΦΗ, αν θέλετε, εν Οπότε καλό είναι να αλληλοσυμπληρωθούμε. συμπληρωθούμε. Επίσης ε, θα συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα με τα γραφεία στα κράτη-μέλη, τα οποία θα συνεργαστούν με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Επιτόπου και με τα διάφορα contact centers, δηλαδή έχουμε αρκετές δομές ε, επικοινωνίας που θα κινητοποιήσουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση και τις επιτόπου εργασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την νεολαία, του εργαζομένου κτλ. Να σας πω ότι είμαστε σε επαφή και με τις διάφορες γενικές διευθύνσεις ε, που έχουν ε, τακτικές επαφές με τις διαφορετικές κατηγορίες πολιτών για να προβούμε σε κάποιες κοινέ δράσεις. Μιλήσατε για την νεολαία σε κίνηση. Πράγματι θα έχουμε κάποιες κοινέ δράσεις ε, διότι σίγουρα αν έχουμε συνέργειες θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερα καλύτερα αποτελέσματα από ότι με δράσεις που θα είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Θα κινητοποιήσουμε και προγράμματα όπως αυτό της Ευρώπης για τους πολίτες με στόχο την συμμετοχή των πολιτών, την προσέγγιση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στον πολίτη μέσω αδελφοποιήσεων και συγκεκριμένων σχεδίων και προγραμμάτων επιτόπου. Στο πλαίσιο λοιπόν και αυτού του προγράμματος θα δώσουμε έμφαση στο Ευρωπαϊκό Έτος ε, για τους ε, πολίτες και για να υπάρξουν πραγματικές συνέργειες. Επίσης ε, μιλήσαμε για τον προπολογισμό. Δεν είναι υψηλός ο προπολογισμό πράγματι. Ελπίζουμε όμως αυτό να αντισταθμιστεί με τις συνέργειες που θα έχουμε και έτσι να έχουμε πολύ μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη. Το τελευταίο ερώτημα αφορούσε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για τις συγκεκριμένες εκστρατείες. Όταν αποφασιστεί ε, πώς θα προχωρήσουμε και όταν έχουμε καταλήξει συμφωνία και μαζί σας και με το Συμβούλιο για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το ευρωπαϊκό έτος, τότε θα εκπονήσουμε και ένα πολύ πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα υποβάλουμε στο Σώμα των Επιτρόπων. Είπατε επίση αν αξιολογούνται οι διάφορε εκστρατείε. Πράγματι, για την ε, εκστρατεία 2013 θα γίνει αξιολόγηση και για τις προηγούμενες χρονιές έχει γίνει αξιολόγηση. Ευρωπαϊκό Έτος Αθελοντισμού μόλις ολοκληρώνουμε τη σχετική αξιολόγηση. Μπορώ να σας δώσω αν θέλετε παραδείγματα. Μπορούμε πάντως να θέσουμε υπόψη σας τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των εκστρατιών. Το ευρωπαϊκό έτος ε, ίσως ε, έδωσε κάποια προβολή σε συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά μετά αυτά όλα συζητήθηκαν και συζητούνται με φορείς ε, και στα διάφορα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό και για το 2011 το ίδιο έγινε γιατί θέλαμε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των εθελοντών, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες και τα προσόντα που αποκτήθηκαν Γενικώ συνεργαζόμαστε με τις γενικές διευθύνσει για να έχουμε συγκεκριμένες και νομοθετικέ ε, τέλος ε, του έτους και όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ολοκληρώνω εδώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν η πρώτη στο τελος του ετους και οπως γινεται καθε χρονο Οδοκληρώνω απόψεων. Ο κύριος Αλαβράκος ξαναζήτησε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους για την τοποθέτηση την οποία κάνανε και πραγματικά παρακαλώ να με υποβοηθήσουν με τις ωραίες σκέψεις τις οποίες εξέφρασα. Ε, βεβαίως ως προς το θέμα της περιφερειακής προβολής ε, το οποίο έθεσε ο κύριος Γιάρ ε, είχα την εντύπωση και επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή ότι θα διοργανωθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πλήθος εκδηλώσεων σχετικά. Αλλά από την άλλη πλευρά ε, εκφράζω και εγώ την άποψη του ότι ο προπολογισμό είναι πολύ λίγος για να μπορέσουμε να δώσουμε την αντίστοιχη προβολή στο ε, επιδιωκόμενο θέμα. Ε, θέλω να σας πω το εξής. σήμερα ήταν μια συζήτηση υγείας, διότι εγώ ήρθα άρρωστος από την Ελλάδα μετά τις γιορτές. Και ήρθα άρρωστος από την Ελλάδα διότι το μόνο το οποίο άκουγα ήταν για την κρίση του χρέους, τα σκάνδαλα, τη, τη διαφθορά, το τι είπε η κυρία Μέρκελ, το τι είπε η κυρία Σαρκοζή, το τι γίνεται στην Ισπανία, το τι γίνεται. Υπάρχουν όμως πέρα από την οικονομία και ορισμένα άλλα πράγματα με τα οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, και πιστεύω ότι οι παλιότερες γενιές που είχαμε λιγότερα χρήματα ζήσαμε με μεγαλύτερη ευτυχία διότι αγαπάγαμε ε, δεν επιδιώκαμε αυτά τα οποία επιδιώκουν οι νεότερες γενιές και βλέπω ότι τους φτιάχνουμε αυτά τα χαρτιά αυτές τις εκθέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα τις βοηθήσουν, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους εκείνους που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Λέμε θα τους εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις να βρουν δουλειά, αλλά δουλειά δεν έχουν. Στην Ελλάδα πήγα και είπα ότι κάντε υπομονή. Ε, σε μια τηλεόραση που μιλούσα δέχτηκα περίπου τα 70 τηλεφωνήματα ότι εντάξει να κάνουμε υπομονή αλλά δεν έχουμε να πάρουμε στα παιδιά μας φαγητό για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όαση να συζητάμε, είναι πολύ ευχάριστο να συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως τα ζούμε ο καθένας στη χώρα του και με τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Και επειδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ίσως θα πρέπει να τα δούμε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα και πέραν του γεγονότος ότι θα εξασφαλίσουμε το σύστημα Solvit, το σύστημα Eures, είναι να, να βρούμε δουλειά στην Ευρώπη και εκεί το βλέπω λίγο δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, ε, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Την ξεκινήσαμε νομίζω με, με καλές ιδέες διότι είναι καλό να ξεκινάμε τη χρονιά μας ε, μακριά από τα ελλείμματα και μακριά από αυτά τα οποία η κυρία Μέλκερ και ο κύριος Σαρκοζή αποφασίζουν και εύχομαι σε όλους σας υγεία και καλή χρονιά. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σαλαβράκου για την παρέμβασή σας. Επομένως κλείνουμε το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Θα δούμε τα σημεία 10 και 11. Ανταλλαγή απόψεων λοιπόν για τις δύο διερευνητικές επισκέψεις ε, στην ε, Γερμανία και στη Ρουμανία. Θα μιλήσουμε πρώτα για την ε, γερμανική επίσκεψη. Η συνάδελφος Γιώτοβα θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω όλοι όσοι λάβαν ε, μέρος αυτή την επίσκεψη στο Βερολίνο να έχουν λάβει τα έγγραφα που εκπονήσαμε. Η επίσκεψή μας στο Βερολίνο αφορούσε ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα και συγκεκριμένα τις υπηρεσίε νεολαίας ε, στη Γερμανία, το έργο τους. Στις 24 Νοεμβρίου 2011 η Επιτροπή Αναφορών ε, οργάνωσε λοιπόν τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο καθότι είχαμε λάβει πολλές αναφορές σε σχέση με το Jugendamt είναι η δεύτερη αποστολή, η δεύτερη επίσκεψη στο Βερολίνο σε σχέση με το θέμα αυτό. Η πρώτη επίσκεψη λάβει χώρα το 2011. Ο κύριος Λυπίσκη, τότε πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Αναφορών, είχε εκπονήσει έκθεση. Έκλεισαν οι σχετικές αναφορές, ε, αλλά έκτοτε λάβαμε πολλές νέες αναφορές για το ίδιο θέμα. Και ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών είναι ακριβώς αυτός, να λαμβάνει τις καταγγελίες που ε, μπορεί να θέλουν οι πολίτες να θέσουν υπόψη μας. Συζητήσαμε λοιπόν τα όλα θέματα που έχουν να κάνουν με την παραβίαση δικαιωμάτων. Τα προβλήματα αυτά δεν πρέπει να αγνοούνται. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσουμε εμείς ε, το δικαστικό σύστημα. Στόχος μας με τη δρυμτική επίσκεψη ήταν να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Και θέλαμε να ακούσουμε τους πάντες οι δυνατόν. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους Γερμανούς συναδέλφους γιατί μας βοήθησαν μας βοήθησαν πάρα πολύ στην διοργάνωση τη επίσκεψη αυτή και μας έδωσαν και πολλές προτάσεις ε, για την κατάρτιση του προγράμματος της επίσκεψης. Προσπαθήσαμε να δούμε γενικά, να προσεγγίσουμε γενικά το ζήτημα και να διατυπώσουμε προτάσεις. Οι αναφέροντες πιστεύουν ότι οι πήκοοι τρίτων χωρών και συγκεκριμένα τα άρθρα 6, 14 και 8 τη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ε, τα άτομα λοιπόν από τρίτες χώρες υφίστανται ε, είναι θύματα παραβιάσεων των δικαιωμάτων με βάση αυτά τα άρθρα. Εμείς στην επίσκεψή μας θελήσαμε να διερευνήσουμε την κατάσταση με βάση τις περιλήψεις των αναφορών που είχαμε λάβει και να δούμε κατά πόσο μας είχαν διαφύγει κάποια ζητήματα. Επομένως, ζητήσαμε τους αναφέροντες να μας πούν ε, αν υπάρχουν ε, προβλήματα τα οποία δεν έχουμε λάβει υπόψη μας. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι το ε, Jugendamt, δηλαδή Γερμανική Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παιδών και Νέων, παρεμβαίνει ε, σε κάποιες περιπτώσεις τα διαζύγια όταν έχουμε μεικτό γάμο. Στόχος βέβαια είναι να προστατευτούν πιο πολύ ε, τα παιδιά και να αποτραπούν ε, ενδεχόμενα απαγωγών και κακομεταχείρισης, κακοποίησης των παιδιών. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 30%, έχει να κάνει, όπως είπαμε, διεθνείς, με μικτούς γάμους. Μετά λοιπόν από την εξέταση των ε, περιπτώσεων, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν έχει αλλάξει τον τρόπο εργασίας ε, της αυτή γερμανική υπηρεσία από το 2006 και μετά. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα που μας απασχόλησε. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα ήταν σε ποιο βαθμό οι γερμανικές υπηρεσίες ε, δίνονται να αξιολογήσουν την αντικειμενικότητα των αποφάσεών τους. Χρησιμοποιούνται μεταφραστές. Και τελικά είδαμε ότι οι περισσότερες αναφορές για τέτοιου είδους προβλήματα έρχονται από τη Γερμανία. Συζητήσαμε και με του συναδέλφου μα από την Επιτροπή Αναφορών τη Bundestag και μας είπαν ότι αυτά τα θέματα δεν τα συζητούν ιδιαίτερα. Α, γιατί είναι θέματα που ανήκουν εμπίπτω στην αρμοδιότητα των τοπικών κοινοβουλίων και όχι του Ομοσπονδιακού. Βέβαια, ε, παρόλα αυτά, 25 αναφορές ε, έφτασαν και μέχρι το Ομοσπονδιακό επίπεδο και επιλήφθηκαν αυτόν οι συνάδελφοί μας. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Jugendamt, ιδρύθηκε το 1922. στα πλαίσια της τοπικής διακυβέρνησης. Може да се съобрази, може и да не се съобрази с това становище τα δικαστήρια τα οποία χειρίζονται τις οικογενειακές υποθέσεις, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου είναι τα αρμόδια για να επιλύσουν τις διαφορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν έχουμε διαζύγιο, και οι δύο ε, πλευρές δεν θέλουν να λάβουν υπόψη τους τις συστάσεις που μπορεί να διατυπώσει αυτή η γερμανική υπηρεσία, το Jugendamt, δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά έχουν δηλαδή αυτό το δικαίωμα. Αλλά αν κρίνει το Jugendamt ότι κινδυνεύει το παιδί ίσως ε, να υποστεί κακοποίηση, ότι υπάρχουν ενδείξεις για υπόνοιε για συμπεριφορά, για απαγωγή κτλ, εκεί μπορεί να παρέμβει. Υπήρξε ο ισχυρισμό ότι οι αποφάσει λαμβάνονται με πολύ υποκειμενικό τρόπο, στηριζόμενε πάνω σε πολύ υποκειμενική βάση. Οι συνάδελφοί μου έθεσαν πολλά ερωτήματα για πάρα πολλά ζητήματα, χωρίς όμως τελικά να καταφέρουμε να συλλέξουμε παρκεί πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται η υπηρεσία. Πώς οργανώνεται. Ουσιαστικά η υπηρεσία έχει περισσότερη σχέση με τις τοπικές κυβερνήσεις, άρα δεν μπορέσαμε να λάβουμε πολλές πληροφορίες από το κεντρικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιβολή κυρώσεων για διοικητικά σφάλματα, πάλι δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο αρμόδιος. Ή ο αρμόδιος φορέας, ή ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας στον οποίο μπορούν να αποταθούν ε, οι γονείς εάν κρίνουν ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Πολλές φορές οι γονείς αναγκάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας να μιλήσουν γερμανικά. Και το έθιξαν αυτό το θέμα οι αναφέροντες. Δεν μπορούν δηλαδή να μιλήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Η επίσκεψή μας όπως είπα, δεν είχε κανένα σκοπό να αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις ε, της Γερμανίας. Αυτό που θέλαμε ήταν να συγκεντρώσουμε πληροφορίες. Ήταν διερευνητική η επίσκεψή μας. Επομένως, ουδέποτε προβήκαμε σε αξιολογήσεις, κρίσεις. Ε, κάποιες φορές, βέβαια, ε, έχουμε κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο τονίσαμε επανειλημμένως ήταν πόσο σημαντικό θεωρούμε να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη τα στοιχεία και οι διατάξεις της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως ε, καλό θα ήταν να έχουμε εδώ ε, μια ομάδα εργασία, ανεπίσημη, ε, μια ομάδα εργασία λοιπόν στην Επιτροπή μας, η οποία θα επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαζύγια. Αυτό είναι μια πρόταση που κάνω ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μου. Να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με του αναφέροντε. Αν και σε άλλε επισκέψει μπορούσε να γίνει αυτό. Σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν εφικτό. Σα ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Ο κύριος Μπουλάν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Όντως, αυτή η διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο ήταν ε, η δεύτερη της Επιτροπής μας. Μετά από την πρώτη επίσκεψη για το πρόβλημα του Jugendamt, ε, ο αρμόδιος ε, διαμεσολαβητής για θέματα οικογενειακά αναγνώρισε προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Γιάρ και Βίλαντ για την ε, οργάνωση αυτής της διερευνητικής επίσκεψης που ήταν άψογη παρόλο που τελικά δεν κατάφεραν να επισκεφτώ την πύλη του Βραδεμβούργου. Εν πάση περιπτώσει, η επίσκεψη νομίζω ήταν πολύ πετυχημένη και αποτελεσματική και ε, διαπιστώνω ότι ε, σήμερα ήταν πολύ πιο ήπια τα σχόλια της κυρίας Γιώτοβα σε σχέση με τα σχετικά σκληρά και μάλλον άδικα σχόλια που απευθύνατε απέναντι στους συνομιλητές μας στη Γερμανία. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον το έργο της αποστολής. Είχαμε πολλούς ε, ε, προσώπους και του Bundestag και του Jugendamt ε, μιλήσαμε και με δικηγόρους και νομίζω ότι λάβαμε γνώση και της λειτουργίας του Jugendamt αλλά και των δυσλειτουργιών που υπάρχουν και αντιμετωπίζονται πολλές φορές. Μπορεί να μην λάβαμε απάντηση σε, όλα, σε όλες τις απορίες μας, αλλά νομίζω ότι προχωρήσαμε αρκετά. Το γερμανικό σύστημα προβλέπει ένα γραφείο προστασίας των νέων. Και είναι σημαντικό γιατί η προτεραιότητα του γραφείου αυτού είναι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων. Πολύ αξιόλογο και αξιέπαινο αυτό το έργο. Είπαμε όμως όταν φτάσαμε στο Βερολίνο ότι δεν ε, ερχόμαστε εδώ ως ε, κριτές, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε γιατί έχουμε τόσες πολλές αναφορές κατά του Jugendamt στην Επιτροπή μας. Και επίσης ε, πολλές φορές δεν ικανοποιούνται οι αναφορές, δεν ικανοποιούνται οι αναφερόμενοι. Ε, αυτοί ήταν η προβληματισμοί. Γιατί δεν δόθηκε συνέχεια και γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Φαίνεται ότι ε, από την επίσκεψη τουλάχιστον φάνηκε ότι και οι υποθέσει που χειρίζεται το Γιούγκεταμ και οι υποθέσει που χειρίζονται τα δικαστήρια αρμόδια για οικογενειακά ζητήματα ε, διεξάγονται με άψογο τρόπο. Και τελικά είναι πολύ μικρός ο αριθμός των προβληματικών περιπτώσεων του Jugendamt. Και φαίνεται ότι υπήρχε μια διαφορά μεταξύ των εξηγήσεων που λάβαμε και των συγκεκριμένων υποθέσεων που παρουσίαζαν δυσλειτουργίες και προβλήματα. Τώρα, ως προς το ερώτημα, ποιος ελέγχει το Jugendamt, Νομίζω ότι ε, μέχρι σήμερα μπορούμε να απαντήσουμε ότι κανένα δεν ελέγχει το Jugendamt. Ε, υπάρχει μερικές φορές δυνατότητα άσκηση προσφυγής για όσους θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν σε ό,τι αφορά το διαζύγιο ή την επιμέλεια παιδιών σε ε, ζευγάρια διαφορετικών υπηκοτήτων, ένας Γερμανός και ένας Αλλοδαπός, ενός Γερμανού και ενός Αλλοδαπού υπηκόου. Και υπάρχει δυνατότητα μέσω προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο, αλλά υπάρχει και δυνατότητα αρμόδιου του Jugendamt να καταγγείλει ε, συμπεριφορά του Jugendamt. Πάντως, διαπιστώσαμε ότι δεν, ασκήθη, δεν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής προσφυγές. Άλλωστε, το Jugendamt δεν είναι ομόσπονδη ή εθνική αρχή, είναι μια δομή που υπάρχει σε κάθε πόλη ουσιαστικά ή σε κάθε αστική περιοχή. Υπάρχουν τόσα Γιούγκενταμ όσο και πόλεις ή περιοχές ε, ευρύτερες αστικές. Είναι μεγάλος ο αριθμός λοιπόν αυτών των Γιούγκενταμ, αυτών των δομών. Και είναι λογικό ότι όταν υπάρχουν τόσες, τέτοια πληθώρα δομών, φυσιολογικό είναι να υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν ασκούν όλοι το έργο τους με τον ίδιο αποτελεσματικό και άμετο τρόπο. Και σε θέματα που αφορούν ε, ζητήματα οικογενειακού δικαίου, ε, διαζυγίου, επώδυνου διαζυγίου μερικές φορές, επιμέλεια ε, παιδιών κτλ. Όλα αυτά τα θέματα έχουν πολύ συγκινησιακά φορτισμένο χαρακτήρα και πολλές φορές και επώδυνο. Πάντως, ε, πρέπει να βρεθεί μια λύση για όσους θεωρούν ότι παραβιάζουν τα δικαιώματά τους ε, που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Πάντως ε, διαπιστώσαμε ότι μερικές φορές καθημερινά έχουμε, λαμβάνουμε στα γραφεία μας καταγγελίες ή αιτήματα ως προς το Jugendamt. Καθημερινά έχουμε μία έως τέσσερις αιτήσει. Βέβαια, φυσικά πρέπει να κάνω μία ανάλυση για να δούμε αν είναι παραδεκτές αυτές οι αιτήσει, οι καταγγελίες, οι αναφορές. Πάντως, είναι μία κατάσταση που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Κατάσταση παραπώνων κατά του Γιούγκενταμ. Με μερικές φορές ένα ζευγάρι χωρίζει και συμφωνούν ε, οι δύο σύντροφοι για τα δικαιώματα επιμέλειας ή επισκέψεων. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα διακανονισμού. Αλλά αν επιδεινωθεί η κατάσταση μεταξύ των δύο συντρόφων, ένας είναι αλλοδαπο και ο αλλοδαπό ε, στη διάρκεια του δικαιώματος επίσκεψης ε, παίρνει το παιδί στην πατρίδα του και στο μεταξύ επιδεινώνονται οι σχέσεις των δύο συντρόφων, είναι πολύ εύκολο ο Γερμανός υπήκος να προσφύγει στο Γιουγκεντάμ και επικαλούμενος κίνδυνο απαγωγής να κινητοποιήσει αυτόν τον μηχανισμό προκειμένου να περιοριστούν τα δικαιώματα επίσκεψης του αλλοδαπού συζύγου. Και να παραμείνει το παιδί στον Γερμανό υπήκο χωρίς καν να υπάρχει απόδειξη απαγωγής. Με απλή υπόνοια του Γερμανού υπηκόου, του Γερμανού συζύγου, μπορεί να στερηθεί ο αλλοδαπός σύζυγος το δικαίωμα επίσκεψης. Και είναι ανυπεράσπιστος ο αλλοδαπός υπηκός απέναντι σε αυτό το μηχανισμό, που είναι χρονοβόρος, ε, δαπανηρός από οικονομική άποψη και ο αλλοδαπός πραγματικά σύζυγος δεν έχει καν δυνατότητα προσφυγής σε μεγάλο βαθμό κατά των αποφάσεων του Γιούγκενταμ. Και ο χρόνος περνάει Προσπαθούμε όμως ε, να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις ε, αντιπαράθεσης μεταξύ δύο συζύγων για υποθετική, για κίνδυνο απλώς απαγωγής, υπόνοια κίνδυνο απαγωγής, λέγοντας ε, στον γονέα μερικές φορές που έχει χρόνια με το παιδί του ότι η συνάντηση θα είναι σοκ για το παιδί, μεγάλος κλονισμός και μερικές φορές παίρνει χρόνια ολόκληρα μέχρι ότου ο ειλικρινής και αφελής ε, ε, αλλοδαπός σύζυγος να ξαναβρει και να ξαναδεί το παιδί του. Σας αναφέρω τώρα μία υπόθεση που είναι συχνή, όχι για όλες τις υποθέσεις που, επιλαβα, που χειρίζεται το Jugendamt, αλλά για τις υποθέσεις που φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη μορφή της αναφοράς. Αυτό το χαρακτήρα συνήθως έχουν οι καταγγελίες που λαμβάνουμε εμείς. Ε, αυτά ως προς τις α, ε, κατεπήγουσες διαδικασίες που εφαρμόζει το Jugendam και που εκφεύγουν οποιοδήποτε ελέγχου. Δεν ε, μπορεί να τεκμηριωθεί η, το βάσιμο αυτής της υπόνοιας απαγωγής που επικαλείται ο Γερμανός σύζυγος. Κάτι που αφήνει διάπλατα ανοιχτή την πόρτα για παρεκτροπές. Και υπάρχουν κάποιες ακραίες οργανώσεις με πολύ εξτρεμιστικές θέσεις και φυσικά δεν τις υποστηρίζουμε που υποδέχονται αυτές τις απελπισμένες, απεγνωσμένες οικογένειες και ε, τις παροτρύνουν μερικές φορές, παροτρύνουν τους αλλοδαποσύζυγους να απαγάγουν τα παιδιά τους και κανονικά τέτοιου είδους οργανώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά ακριβώ λόγω του πλαισίου αθούν όλο και περισσότερο τέτοιου είδους εξτρεμιστικές οργανώσεις. Βέβαια, Έχουμε και την περίπτωση της Συμφωνίας Βρυξελών 2α. Υπάρχουν κάποια δικαιώματα με βάση το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει το δικαίωμα ε, προσφυγής κατά δράσης από υπάλληλο. Επίσης, μερικές φορές υπάρχουν διακριτικές ε, μεταχειρήσεις ε, για τη χρήση της μητρικής γλώσσας, ε, δικαίωμα για δίκαιη δίκη και ενημέρωση το συντομότερο δυνατό, δικαίωμα χρηστής διοίκησης ή δικαίωμα κρόασης, ώστε να εξασφαλίσετε πρόσβαση στη δικογραφία και τα δικαιώματα φυσικά των παιδιών. Όλα αυτά τα δικαιώματα, στις αναφορές που εξετάσαμε στην Επιτροπή μας τουλάχιστον, φαίνεται ότι δεν γίνονται σεβαστά, δεν τηρούνται. Και αυτές οι επικρίσεις δεν ασκούνται μόνο από εμά, ακόμη και στη Γερμανία. Βλέπουμε σε γερμανικές εφημερίδες ε, αρνητικά σχόλια και κριτική κατά του Ιούγκεντα. Οπότε βλέπετε το πρόβλημα ε, επισημαίνεται ακόμη και στην ε, χώρα προέλευσης του στη Γερμανία. Εγώ χαίρομαι πάντως που πραγματοποιήσαμε αυτή τη δεύτερη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο και μετά τις συνομιλίες που είχαμε ε, το Υπουργείο Αρμόδιο για Οικογενειακά Θέματα έδειξε προθυμία για συνομιλίες μαζί μας, θα πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να παραπέμψουμε στο Υπουργείο αυτό τις 4-5 χαρακτηριστικές υποθέσεις με καταγγελίες κατά του Ιούγενταμ που είναι πραγματικά υποθέσεις που καταστρατηγούν ε, κατάφορα τα δικαιώματα των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε σε αυτό το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα οικογένειας, ε, ζητώντας σε έφθετο χρόνο να διευθετήσει αυτά τα προβλήματα και θα δούμε τότε αν μέσω του αρμόδιου Υπουργείου μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους αναφερόμενους. Ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν και άλλες λύσεις. Πάντως, ε, τα ε, περισσότερες αιτήσει που λάβαμε και αυτές που καθημερινά λαμβάνουμε, αιτήσει ε, αναφορές καταγγελίες στα γραφεία μας, είναι πραγματικά ανησυχητικές. Θεωρώ ότι υπάρχει διαρθρωτικό πρόβλημα στη Γερμανία. Δεν θέλω φυσικά να επέμβω σε εσωτερικά θέματα διοργάνωσης στη, Γερμανία και ε, δομής των διαφόρων ε, γραφείων. Θα ήταν άτοπο κάτι τέτοιο. Αλλά καλό θα ήταν ε, ίσως να υπάρχει ένας ε, διαμεσολαβητής σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατηδίων. Γιατί αν είχαμε ένα συνομιλητή που θα μπορούσε στη συνέχεια να παραπέμψει το θέμα στον Ομοσπονδιακό Διαμεσολαβητή ή αυτός να έχει συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές, νομίζω ότι η λύση στο πρόβλημα θα ήταν πολύ πιο άμεση και ταχεία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα στη λειτουργία του Jugendamt και στα δικαστήρια, αλλά μέσω ενός τέτοιου διαμεσολαβητή θα μπορούσαμε να τα διευθετήσουμε πιο γρήγορα. Για να σταματήσει αυτός ο καταιγισμός ε, των αναφορών από τη Γερμανία κάτω του Jugendamt. Πιστεύω θα πρέπει να γίνει αυτή η προσφυγή κατά της Γερμανίας. Αντιλαμβάνομαι ότι μακρηγόρησα, πάντως ε, πολύ συχνά διαπιστώνω ότι ζητούμε από τους αναφερόμενους να ασκήσουν προσφυγή κατά το οργάνου που έλαβε την απόφαση. Κάτι τέτοιο όμως αντιβαίνει στο ίδιο, στην ίδια τη φύση του ένδικου μέσου, του μέσου προσφυγής. Δεν μπορεί κάποιος να είναι και, δι, και δικαστής ε, και κατηγορούμενος. Θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη, άλλη δομή στην οποία θα πρέπει να απευθυνθεί για να προσβάλλει μια τέτοια πράξη ο αναφερόμενος, ε, ο θυγόμενος. Ελπίζω το αρμόδιο Υπουργείο της Γερμανίας να μας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και ευελπιστώ ότι θα βρει η Γερμανία λύσεις για τα προβλήματα αυτά για να μην φτάνουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλαντ έχει το λόγο τώρα. Ähm, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Γιώργο. που που με την στάση του και αυτό συνέβαλε στην επιτυχία αυτής της ε, επισκέψεως. Ως ε, νομικός, στην προηγούμενη αυτοδρομία, φρόντισα να έρθω σε επαφή και με την ε, οικογένεια και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα και από τη δουλειά της ESD και των, και των αρμοδίων για την επικοινωνία με το δικαστικό σύστημα. Είδαμε λοιπόν τι κάνουν οι δικαστές, είδαμε ότι υπάρχει προσπάθεια για αντιμετώπιση των υπερσυνοριακών προβλημάτων και η προσπάθεια μέσω του ESD να ε, διευρυνθεί ενημέρωση για το πλέγμα διατάξεων που ισχύει σε άλλο κράτος. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η επίσκεψη. Αλλά κατέστη πάνω απ' όλα η δεύτερη αυτή ε, επίσκεψη απαραίτητη γιατί δεν είχε ικανοποιητικά διεξαχθεί η πρώτη. Δεν είχαμε δηλαδή φροντίσει επαρκώς με αρκετή προετοιμασία να οργανώσουμε την πρώτη επίσκεψη. Είχαμε μόνο ένα έγγραφο ε, εργασίας στο οποίο καταγραφόταν μόνο η επίσημη θέση ε, και ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως είχαν. Γι' αυτό κατέστη απαραίτητη η δεύτερη επίσκεψη και όχι γιατί είναι τόσο τεράστια τα προβλήματα και δεδομένε οι παραβάσει στη Γερμανία. Και δεν θέλω να καταστήσω κάτι σαφές όταν μιλούμε για σατανικές μηχανές και θα ήθελα να διορθώσω τον συνάδελφο από τη Γαλλία. Όταν λένε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ξέρω αν ε, οι εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε σε άλλη γλώσσα ακούγονται κάπως παράξενα, αλλά πάντως είναι εκφράσεις που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον εσκεμμένος Άλλο να πούμε δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, άλλο δεν είναι πλήρηση προστασία τους, που συμβαίνει σε κάθε κράτος μέλος, Α κοιτάξουμε τη ε, νομολογία και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά το να λέμε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ε, αγνοούνται ε, συστηματικά είναι πάρα πολύ βαρύ. Υπάρχει συστηματική καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν, σε ένα κράτο των 80 εκατομμυρίων, όπω η Γερμανία, είναι πιθανόν να υπάρξουν κάποια προβλήματα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες διαζυγίων. Είναι τη χιλίες τα ποσοστά στα οποία μπορεί να προκύψει κάποια δυσκολία. Και αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι αντιμετωπίζεται έξω από το ε, δικαϊκό σύστημα ή το δικαστικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να προσφύγει σε ένα δικαστήριο. Ας κοιτάξουμε πόσο διαρκούν σε κάποια κρατημέλη, στα επιμέρους κρατημέλη, οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων. Στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια κράτος του Νότου, όχι της Γαλλίας, λέγεται, λέγεται ότι εάν είναι, ε, ότι είναι τόσο μακρές οι διαδικασίες των δικαστηρίων, όπου εάν το ζευγάρι είναι μεικτό, με γερμανό υπήκο το ένα μέλος του, προτιμά να πάνε στη Γερμανία να στήσουν διαζύγιο παρά να περιμένουν στο κράτος αυτό την έκδοση αποφάσεως. Γι' αυτό λοιπόν τώρα αν έχουμε μια υπηρεσία κοινωνική η οποία δεν ε, φρόντισε εγκαίρω τα δικαιώματα του παιδιού κτλ. είναι ένα ποστό επί της χιλής όπως είπα. Η δε εναλλακτική είναι η περίπτωση Κολόμπο. Η εναλλακτική είναι η υπόθεση Κολόμπο, δηλαδή η περίπτωση απαγωγής του παιδιού και άρνηση κάθε νομικής προστασίας, παράβαση κάθε έννοιας ε, νόμου και δικαίου απαγωγή του σε τρίτο κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με κανένα δικαίωμα επίσκεψης και επικοινωνίας με το παιδί, δηλαδή δράση εγκληματική που εν τέλει και στην περίπτωση Κολόμπο στην Ιταλία συγκεκριμένα ο εμπλεκόμενος γονέας κατέληξε στη φυλακή. Διότι ήταν περίπτωση απαγωγής τέκνου. Επομένως αυτή είναι εναλλακτική έναντι μιας δικαιοδοσίας η οποία ενδεχομένω βραδιπορεί. Και ναι, ομολογώ ότι διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε παράπονα για κάποια προβλήματα στις κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προστασία ανηλίκων. Αυτά τα βλέπουμε τακτικά σε όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Το ότι έχουμε τώρα μία, το ότι λέγεται μάλλον ότι υπάρχει μια πληθώρα, ε, μια πλημμυρής πλημμυριση υποθεσεων τέτοιων ε, στη Γερμανία, νομίζω ότι είναι πολύ άδικο. Και πρέπει επίση να επισημάνω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει καριέρα εγκληματική σταδιοδρομία με το να αναλαμβάνουν απαγωγέ τέκνων σε περιπτώσει τέτοιων μεικτών διαζυγίων και προσφέρουν τι υπηρεσίε του στον ενδιαφερόμενο γονέα. Άρα λοιπόν, το ποιο είναι αυτό ο οποίο κινεί τα νήματα, ίσω θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και ίσως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όταν ε, φτάνουν με διαδικασία μη συνενετική οι υποθέσεις αυτές στα δικαστήρια, όταν είναι δηλαδή με αντιπαράθεση διαδικασίας αυτές, η απόφαση του δικαστηρίου μοιραία θα φανεί άδικη στον έναν από τους δύο τα δύο μέρη, θα θεωρήσει ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Και εάν δεν υπάρχουν άλλε ε, διασφαλιστικέ δικλείδε, υπάρχει ο κίνδυνο να περιέλθει σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα που θα πρέπει να κοιτάξουμε, ότι έχουμε να κάνουμε με ευρωπαϊκό δίκαιο, Γερμανού γονεί, Γερμανού υπηκόου στα παιδιά του, απευθύνονται στο γερμανικό δικαστήριο, έχουμε κοινωνική υπηρεσία αναλύκων ε, γερμανική και Εδώ θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε να εφαρμόζεται και να, να παρακολουθεί μάλλον την εφαρμογή του δικαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα. Δεν αρκεί δηλαδή το να επισημαίνεται αφηρημένο ότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στην διοίκηση. Και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιο άλλο κράτο του Νότου, στο οποίο ενδεχομένω να ακούγονται κάποιες κατηγορίες πολύ σοβαρέ για την έννοια της ε, υπηκότητας, της ηθαγένειας τη Όλα αυτά νομίζω πρέπει να τα δούμε με μια κάποια απόσταση. Ευχαριστώ πολύ την ε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στο Βερολίνο, λέει ο κ. Μπέκερ. Εχθές ε, ετοίμασα μια, ε, έλαβα μάλλον την έκθεση, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να την διαβάσω με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να πω ότι και, στις, ε, και από τους συναδέλφους Γιάρ και Βίλαντ μπόρεσα να διδαχθώ πολλά στην ε, αποστολή αυτή, η οποία μας επέτρεψε να εξετάσουμε εις βάθος τα ζητήματα και όπου είναι πολύ επικοδομητικός ο ρόλος του των συνομιλητών μας. Πολλά είναι λοιπόν αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και να συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό στη συζήτηση που αναπτύσσεται ευρύτερα. Εκ μέρους όμως Επιτροπής των Αναφορών θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής. Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα γραπτός να καταθέσω κάποιες προτάσεις, γιατί δεν ήμουν έτοιμος να τις διατυπώσω όπως θα ήθελα. Ε, νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάς. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην αντιπροσωπεία που βοήθησε στην ε, διεξαγωγή αυτής της ε, αποστολής. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Βίλαντ με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό μετά όσα είπε. Θα ήθελα πάντως να πω ότι κάποια αισθήματα μείνανε εκρεμή. Η γερμανική πλευρά είχε προτείνει μια μάλλον τεχνική επίσκεψη. Εμείς ως Επιτροπή είπαμε ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό. Επισκεφθήκαμε επί δύο-τρεις μέρες συνεχώς από το ένα μέρος στο άλλο στην περιοχή που είχαμε προβλέψει, κοιτάξαμε ό,τι μπορούσαμε και οποιαδήποτε ενδεχομένως ακόμη ε, ανοιχτά ζητήματα, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, πιστεύω θα μπορούσαμε να τα σημειώσουμε στο τελικό κομμάτι της εκθέσεως και να τα αποστείλουμε στις γερμανικές αρχές για να ζητήσουμε κάποια αντίδραση από πλευρά τους. νομίζω ότι θα ήταν δυνατόν, δεν νομίζω έχει κανεί αμβολία, ότι μπορούμε να αποστείλουμε παρατηρήσει, ερωτήσει στι γερμανικέ αρχέ και να ζητήσουμε απαντήσει. για σε τελευταία ανάλυση, μέσα σε αυτέ τι δύο μέρε που είχαμε την ε, αποστολή, δεν ήταν δυνατόν να καλύψουμε όλα τα θέματα. Μας περιπτώσει, το πεδίο δράσεω τη Υπηρεσία Προστασία Ανηλίκων είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε σε άλλη περίπτωση ζευγάρι μη Γερμανών μεταναστών, εν πάση περιπτώσει, στη Γερμανία, που είχαν επαντρευτεί όμως στη Γερμανία και όπου η μητέρα ζητούσε να προστατευτεί το παιδί, να αφαιρεθεί δηλαδή από την επιτροπή της οικογένειας προκειμένου να το προστατέψει με τον τρόπο αυτό από την βία η συμπεριφορά του πατρός. Άλλες περιπτώσεις όπως αυτή υπάρχουν ε, στην περίπτωση αυτή το, η σχετική κοινωνική υπηρεσία αναγνώρισε δίκαιο στο αίτημα της μητέρας και όντως πήρε το παιδί από την οικογένεια με αποτέλεσμα όμως στη συνέχεια ο πατέρας αυτός να βρει την κόρη του στο δρόμο και να τη σκοτώσει με ένα περίστροφο. Ε, Επομένω, εκεί πέρα το ζήτημα που ετέθη ήταν περισσότερο γιατί δεν δόθηκε περισσότερη προστασία στο παιδί αυτό από τη στιγμή που αφαιρέθηκε από τους κόλπους της ε, φυσικής του οικογένειας. Και η ε, επικοινωνία και η ευαισθητοποίηση του πατέρα, γιατί εκείνο θεώρησε μόνο ότι του αφαιρέσαν το παιδί του και ότι είχε κάθε δικαίωμα πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, μπορεί κάποτε τα διαζύγια να διεξάγονται κατά τρόπο ήρεμο προς τον προσδορισμό της γονικής μέρημνας και της φροντίδας για τα παιδιά ή ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει, αλλά όχι πάντα. Και τότε που ξεκινάνε τα προβλήματα. Ε, μόνο και μόνο από το γεγονό ότι ο ένα γονιό μένει στο ένα μέρο και ένα στο άλλο, ο πατέρα στο μόναχο και η μητέρα στη Σικελία, φερειπίν μετά το διαζύγιο, το παιδί αναγκάζεται να πηγαίνει πότε στον έναν και πότε στον άλλον. Ε, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται με ευαισθησία και να κρίνονται μέσα στο πλαίσιο βεβαίω του ε, δικαιώματο και τη υποχρέωση για ανατροφή του παιδιού, για εκπαίδευση του παιδιού κτλ. Πάντω, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε με την έκθεση να διατυπώσουμε τα ανοιχτά ακόμα ζητήματα και να περιμένουμε να λάβουμε απαντήσει. Ο κύριο Αλαβράκο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι η αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα καθιδρύεται κατά περίπτωση. Δηλαδή, μπορούμε να επιληφθούμε ενό θέματο μετά από μια αναφορά. Μόνο αυτού του συγκεκριμένου θέματο. Γενικεύσεις δεν μπορούμε να κάνουμε πρέπει να εξετάζουμε το κάθε θέμα που μας τίθεται και να βλέπουμε εάν στο συγκεκριμένο θέμα καθιδρύεται αρμοδιότητα της Επιτροπής μας είτε για παράβαση της κοινωνικής νομοθεσίας είτε για παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, από την εμπειρία μου είμαι κατά των γενικεύσεων διότι ξέρετε η στατιστική η οποία είναι ο καλύτερος ε, δείκτης δείχνει πολλές φορές ότι έχουμε μικρές στατιστικές παραβάσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για τον κάθε έναν που του παραβιάζεται το ανθρώπινο δικαίωμα είναι η μοναδική του περίπτωση. Επομένω, δεν θα συμφωνούσα στη γενίκευση και το χαρακτηρισμό του δικαιακού συστήματο ενό κράτου σαν τη Γερμανία, που να πούμε ότι είναι καλό ή κακό το δικαιακό σύστημα σε σχέση με την αντιμετώπιση των διαζυγίων, των μεικτών γάμων και την ε, ε, παροχή όλων εκείνων των διατάξεων ε, προστασία σε όλες, με όλες εκείνες τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου ή του κληρονομικού δικαίου ή οποιοδήποτε κλάδου δικαίου. Και γι' αυτό θα έλεγα, δεν είδα, δεν είδα την ε, έκθεση της Επιτροπής. Η ένστασή μου επομένως είναι σε σχέση με την περίπτωση που εξέτασε, διότι προφανώς πήγε εκεί και εξέτασε μια, δύο, τρεις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάνει αναφορά. Για μόνο αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να εκφράσουμε απόψε την Επιτροπή νομίζω. Δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Και ε, εν πάση περιπτώσει ίσως θα πρέπει να θέσουμε και τους κανόνες στην Επιτροπή για να διατηρήσουμε και τη σοβαρότητά μας σε τι, τι επιλαμβανόμεθα και τι αποφασίζουμε διότι ήδη νομίζω ότι και για το μέλλον δημιουργούμε ενό είδους ε, νομολογία η οποία πρέπει να είναι ασφαλής και πρέπει να είναι ασφαλής για αυτούς που θα την ακολουθήσουν. Ξέρετε ότι στην Αγγλία δεν υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει το δίκαιο των cases και ε, με τις υποθέσεις αυτές από το 1600 μέχρι τώρα περπατάει το δικαιακό σύστημα της Αγγλίας μια χαρά. Γι' αυτό λοιπόν ε, το θέτω αυτό υπόψη σας και ίσως θα πρέπει να βάλουμε κανόνες πώς βάζουμε τις εκθέσεις μας. Όχι γενικά και αόριστα για τη συγκεκριμένη και μόνον περίπτωση την οποία επιλαμβανόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Ο κύριος Μπουλάν ξαναζήτησε το λόγο, αλλά ξεπερνάμε το χρόνο. Σας παρακαλώ, χρονοφίδο. Μισό λεπτό μόνο, ε, κυρία Πρόεδρε, για τους ε, φίλους και συναδέλφους από τη Γερμανία. Όπως είπε ο κύριος Βίλαν, το θέμα δεν είναι αν είναι σκεμμένη η πολιτική αυτή. Γιατί πριν από λίγο μίλησε για κάποιες εξτρεμιστικές ιδέες κάποιων οργανώσεων και αντιτάχθηκα σε αυτές, γιατί εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το πρωταρχικό ζήτημα και σίγουρα δεν θεωρούμε ότι είναι σκεμμένη αυτή η πολιτική. Αν μη τι άλλο, εξαιτία τη πληθώρα ε, των Jugendamt και της πολύ κατακαιρματισμένης δομής. Αλλά γιατί έχουμε τόσες πολλές αναφορές ε, θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει για να δούμε τι λύση μπορούμε να προσφέρουμε. Τα ε, κολέγα ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σύντομα θα σας δώσω και την τελευταία, την τελική εκδοχή της έκθεσης. Θα παρακαλώ τους συναδέλφους ε, να μου υποβάλουν εγγράφος στα σχολιά τους, ούτως ώστε ό,τι θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να περιληφθεί στην έκθεση να μπορέσω να το συμπεριλάβω. Να κάνω κάποια σχόλια τα οποία θεωρώ σημαντικά σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος ε, Σαλαβράκος. Επειδή δεν ήταν ε, στην αντιπροσωπή αυτή, ίσως έχει μείνει με μία εσφαλμένη εντύπωση για το πόσο είχε οργανωθεί αυτή η επίσκεψη. Δεν επεξεργαστήκαμε μία ή δύο συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι για καμία συγκεκριμένη περίπτωση δεν συζητήσαμε στη διάρκεια τη επίσκεψη. Ε, το είδαμε γενικά το θέμα. Αυτό που κάναμε ήταν ότι ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες ε, υποθέσεις. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τον ε, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο κύριος Αλαβράκος. Δηλαδή δεν μπορούμε με βάση δύο, μία, δύο, τρεις υποθέσεις να καταλήγουμε σε γενικά συμπεράσματα. Επίσης έγινε, μου έγινε μια ερώτηση για τα ποσοστά, τα ποσοτικά δεδομένα. Εδώ θέλω να πω το εξή. Οποιοδήποτε πολίτης έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα και έχει στραφεί σε εμά, πρέπει να ακουστεί. Σε ό,τι αφορά την πρόταση να ζητήσουμε έγγραφες απαντήσεις από τον οργανισμό, θα το λάβω υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σαλαβράκο. Ότι ε, δεν μίλησα ειδικό για την έκθεση. Μίλησα ε, γενικώ για την αρμοδιότητά μας. Δεν μπορούμε να επιλαμβανόμεθα χωρίς αίτηση κάποιου ε, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να λαμβάνουμε αποφάσεις αορίστως. Πρέπει να υπάρχει αίτηση. Χωρίς την αίτηση πρέπει να έχουμε case, πρέπει να έχουμε περίπτωση επί της οποίας θα αποφασίσουμε. Γιατί αλλιώς είμαστε αναρμόδιοι, παραβιάζουμε την αρχή της επικουρικότητας. Μιλάμε για να σταθούμε πολύ σοβαρά πάνω σε αυτή τη δουλειά την οποία κάνουμε και πρέπει για το μέλλον κάθε απόφασή μας και αιτιολογημένη να είναι και να αποτελεί για το μέλλον έναν οδηγό Εάν πάμε ειδικώ και κάνουμε ερωτήματα εμεί δεν δικαιούμαστε, δεν θα εισαγγελεί. δεν θα του κλάδου των εισαγγελέων. θα του, του δικαιοδοτικού κλάδου. Κάποιο προσφεύγει σε εμά και απαντούμε εάν έχει δίκιο ή δεν έχει άδικο με βάση την κοινωνική νομοθεσία. Δεν μπορούμε εμεί αορίστως να πούμε έχει δίκιο μια μερίδα ανθρώπων απροσώπους. Πρέπει να έχουμε case. επομένω, αυτό που είπα δεν το είπα για την έκθεσή σα το είπα σαν γενικό κανόνα πάνω στον οποίο πρέπει να επιλαμβανόμεθα τις περιπτώσεις σαν Επιτροπή. Διότι αλλιώς δεν θα έχει νομικό αποτέλεσμα αυτό το οποίο κάνουμε. Νομίζω ήμουν επαρκή στην εξήγησή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιώτοβα για την εργασία που φέρατε σε πέρας. Ε, να ευχαριστήσω και όλους όσους έλαβαν το λόγο στη συζήτηση αυτή που θεώρησα αρκετά ενδιαφέρουσα. Η συζήτηση άλλωστε που θα συνεχιστεί. Όπως βλέπετε από τη διαδικασία ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Στην ημερήσια διάταξη προβλεπόταν και η συζήτηση της διερμητικής επίσκεψης στη Ρουμανία, αλλά πέρασε η ώρα. Σας παρακαλώ λοιπόν να αναβάλουμε την εξέταση του θέματος αυτού για τη μεσημεριανή μας συνεδρία. Θα το πρώτο θέμα της μεσημεριανής συνεδρίασης, εάν δεν διαφωνείτε.